κάτι το οποίο το αξίζει. Ο κύριος Φούλε τώρα θα αναλάβει την σκητάλη μετά την είπατε εκπρόσωπο για να παρουσιάσει το επόμενο θέμα που αφορά τη στρατηγική για τον εύξηνο πόντο. Όταν πάρει τη θέση του μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Uh, uh, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χαρά μου συζητώ το θέμα αυτό εκ μέρους της ΥΠΑ ΕΕ, της εκπροσώπου και αντιπροέδρου το θέμα αυτό της ε, περιφερειακής συνεργασίας και προπτικές όσον αφορά τη συνεργασία μας με τις χώρες του Ευξήνου Πόντου. Δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό το Κοινοβούλιο. Η περιοχή του Ευξήνου Πόντου είναι μια πολύ πλούσια περιοχή και σε φυσικούς πόρους και σε ανθρώπινους πόρους. Και είναι δίωδος που ενώνει Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή και προσφέρει δυνατότητες να εντοπιστούν τομείς που υπάρχουν κοινά συμφέροντα για συνεργασία. Από το 2007 με προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπλακεί άμεσα στι προσπάθειε καταβάλλοντα στον Πόντο. Υπάρχουν σημαντικέ δυνατότητε και προκλήσει στην περιοχή. Απαιτείται συντονισμό και δράση. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τη συνέργεια για τον έξινο πόντο 2008 είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Καμιά φορά με ρωτούν αν αυτή η συνεργασία των εύξηνο πόντο δεν αλληλεπικαλύπτει την ανατολική εταιρική σχέση. Εγώ απαντώ όχι. Η εταιρική συνεργασία φέρνει πιο κοντά τους ανατολικούς μας εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικής συνεργασίας και οικονομικής ολοκλήρωσης. Η συνεργασία με τις χώρες του Ευξήνου Πόντου φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον Ευξήνο Πόντο, συμβάλλοντας την περιφερειακή συνεργασία. Και τώρα να προσθέσω κάποια προσωπικά σχόλια Βέβαια υπάρχει και διάδραση μεταξύ της ανατολικής συνεργασίας της χώρας ανατολικά της Ευρώπης και με τη συνεργασία με τον έξινο πόντο. Η συνεργασία με τις χώρες ανατολικές έχει γίνει σημαντικό κομμάτι των προσπαθειών μας και δημιουργούνται δυνατότητε επίση για συνεργασία με τι χώρε περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο που θα μα παρέχει τι ανάγκε συνέργειε όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών μα στην περιοχή. Θα συναθρήσουμε τα όσα κάνουμε με τους εταίρους μας θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε σύμπραξη διασυνοριακά και να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο στην περιοχή. Αξιότιμα μέλη. Έχουμε πολλά συμφέροντα, περιβάλλον, θέματα αφορούν τη θάλασσα, αλληλεία, ενέργεια, μεταφορές, ε, μετακίνηση, ασφάλεια. Εμείς εστιαζόμαστε όμαστε σε τρεις τομεακές συνεργασίες, περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια. Τον Μάρτιο του 2010 ξεκίνησε η συνεργασία στον περιβαλλοντικό τομέα. Επιπλέον, έχουμε πρόγραμμα σημαντικό της συνεργικής συνεργασίας στην περιοχή. Ο προπολογισμό για 2007-2013 για το πρόγραμμα του ξύνου σε δεσυνοριακό επίπεδο αυξήθηκε από 17 σε 25 σχεδόν 26 εκατομμύρια ευρώ. 18 προγράμματα εφαρμόστηκαν. Καλύπτονται τις προτεραιότητες. Στην περίοδο 2007-2013. Προγράμματα που αφορούν τον εύξηνο πόντο. Υποστηρίζουμε συνεργασία διασυνοριακή για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Κοινή χρήση των πόρων και γνώσεων για προστασία του περιβάλλοντος και για διαφύλαξη αυτού. Υποστήριξη της παιδείας, πολιτισμικών πτυχών και σχετικών πρωτοβουλειών για να δημιουργηθεί ένα κοινό περιβάλλον πολιτισμικό στην περιοχή του Ευξηνοπόντου. Όμω, δεν προχωρήσαμε όσο θα θέλαμε όσον αφορά αυτέ τι συνεργασίε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξαναεξετάσουμε πώ αυτή η συνεργασία μα στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου μπορεί να προχωρήσει. Καλωσορίζω λοιπόν τη δυνατότητα να το συζητήσω μαζί σα. Όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική των Ευξήνου πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει δεκτή καλά και εντό Ευρωπαϊκής Ενώσεω και μεταξύ των χωρών του Ευξήνου Πόντου που δεν συμμετέχουν στην Ένωσή μα. Εν τω μεταξύ, εμείς πρέπει να δούμε πώς θα αναζωογονήσουμε τη συνεργασία με τις χώρες του Ευξήνου Πόντου εν ώψη μελλοντικών εξελίξεων. Πρέπει να σκεφτούμε τρία πράγματα πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναζωογονήσουμε την προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τη συνεργασία στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη την ποικιλία των σχέσεων που έχουμε με τι χώρε τη περιοχή. τις παρευξήνιες. Έχουμε υποψήφια χώρα την Τουρκία. Στρατηγικότερο έχουμε τη Ρωσία, συν τους εταίρους μας εντός της Ανατολικής Αττικής Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Τζορμπαϊτζάν. Πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη τις καμιά φορά δύσκολες σχέσεις που έχουν αυτές οι χώρες μεταξύ τους ή με γειτονικέ χώρε που είναι γειτονικέ των παρευξηνίων χωρών. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα άλλα πλαίσια συνεργασία στην περιοχή. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Στον τομέα τον περιβαλλοντικό, η Επιτροπή Τευξίνου Πόντου είναι σημαντικό επιτροπη τευξινων ποντου ειναι σημαντικο παραγων και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει να γίνει αποδεκτή σαν πλήρε μέλο. Θέλουμε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για συνεργασία συνεργασία μας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου, μάλιστα από την ευκαιρία της 20ης επαιτίου και της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει στις 26 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Αναζωογωμένη συνεργασία στον Εύξηνο Πόντο και συμμετοχή στους φορείς οικονομικής συνεργασίας του Ευξήνου Πόντου θα δώσει μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας και για να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσίας και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Είναι σημαντική εμπλεκόμενη φορή στην περιοχή και οι δύο. Και τρίτον, σημαντικότερο είναι αυτό το σημείο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες, τα σχηρά σημεία που μας δίνει η συνθήκη της Αβώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε οι εσωτερικές μας πολιτικές και εξωτερικέ εξωτερικές να εφαρμοστούν σωστά και θα είναι πολύτιμες οι ανταλλαγές απόψεων με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Πρέπει να συνεχιστεί ο προβληματισμός μας, να δούμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη σωστή πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι αυτής της σημαντικής περιοχής. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Λέω Πρόεδρο, πρώτο αγορητή είναι ο κ. Ουγγουρεάνου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Έχω ε, συντάξει μια έκθεση όσον αφορά την μεταφράση και σα επιβεβαιώνω ότι έχουν περάσει 15 μήνε από τότε που εμεί ζητήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια κοινοτική στρατηγική σε σχέση με την μαύρη θάλασσα και έτσι να αναβαθμίσουμε την συνέργεια με την περιφέρεια αυτή, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η πολιτική το 2008 είχαμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και τότε που ξεκίνησε η συνέργεια με την Μαύρη Θάλασσα, αυτό εξυπηρέτησε σε πολλά μέτωπα. Ναι, ναι, πρόκειται για μια αυτάρκη αυτόνομη πολιτική και επίσης έτσι έχουμε χαρακτηρίσει την περιοχή ως στρατηγικά σημαντική για την Ένωση. Πέρασαν τέσσερα χρόνια και τώρα τα αποτελέσματα των επιδόσεων μας είναι 7. Γιατί αντί για κάποια πολιτική, η περιφέρεια αυτή είναι κάτι σαν μαύρη τρύπα. Τίποτα δεν έχει γίνει από το 2008. Καμία πολιτική, κανένα έγγραφο στατικής σημασίας για την περιοχή αυτή. Επίση, οι προκλήσει στην περιφέρεια αυτή δεν θα κάθονται να περιμένουν πότε θα κάτσει να στοθεί στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η μαύρη θάλασσα. Είναι μια περιοχή που είναι μπάρο τα αποθήκια όσον αφορά τις εντάσεις, τις συγκρούσεις. Έχουμε θέματα εκεί πέρα ε, για το περιβάλλον, για την πολιτική της θάλασσας. Που δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Οι δύο περιπτώσεις, το 2008 από το και το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να έχουμε αναβάθμιση αυτής της συνέργειες. Ακόμα όμως τα πράγματα έμειναν στάσιμο. Ακόμα περιμένω την Κομισιό να εκπονήσει μια σχετική στρατηγική. Ρούτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Black Sea region, it's a region of strategic importance. As been already mentioned, there are... Πάρα πολύ στρατηγική σημασία είναι αυτή η χώρα, γιατί έχουμε εκεί πέρα μια σειρά χαρών της Ένωσης, Έχουμε υποψήφιους Όπω όπως η Τουρκία. στρατηγικός εντός είναι και η Ρωσία. Αλλά και τους ανθρωπικούς γείτονες οπότε είναι προς το συμφέρον μας να βοηθήσουμε το ώστε εκεί να πρετανεύσει η σταθερότητα, η ευημερία, η ασφάλεια, εκεί η κοινωνικότερη διότι μάλιστα εκεί έχουμε κάποιες συγκρούσεις και όλα αυτά ε, εκκρεμούν και ελοχεύουν για πάρα από 20 χρόνια. Τι θα κάνουμε, νομίζω ότι η αυτή προσέγγιση που ανέφερε ο Επίτροπος ε, έρχεται να συμφωνήσει με κάποιες από τις πολιτικές μας. Με τα, μεταφορά κλπ. Και, και είναι σωστές αυτές τις διότι αν καθίσουν μια ματιά εις το έργο το οποίο έχει επιτελέσει η κοινοβουλευτική συνέλευση, ακριβώς αυτά είναι τα θέματα εις τα οποία έχουμε δραστηριοποιηθεί. Άρα θα πρέπει αυτή την πολιτική να την βοηθήσουν. Θα πρέπει ακριβώς να έχουμε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, τη διασύνδεση των λιμένων. Να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εκεί γειτόνων και βέβαια να βοηθηθεί ο τουρισμός, η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον. Και με αυτόν τον τρόπο βήμα-βήμα να βοηθήσουμε να αναζητηθούν κάποιες λύσεις ή σε αυτές τις προστιβές, τις συγκρούσεις, τις διαφορές. Επομένως, η προσέγγιση που μας εξήγησε ο Επίτροπος είναι ορθή. Να συμφωνήσουμε μαζί του, να είμαστε πιο δυναμικοί σε σχέση με αυτή την συνεργασία Μέλτζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τον τελευταίο καιρό σίγουρα έγιναν αρκετά πράγματα ώστε να ενισχυθεί η ανατολική εταιρική σχέση και να γίνει πιο αποτελεσματική. Τα κίνητρα για περισσότερα είναι σίγουρα ως προσέγγιση, σωστή προσέγγιση, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες αλλαγές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα φυσικά για τις χώρες στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι κινητήρας προς αυτήν την κατεύθυνση. Η περιφέρεια περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας θα κερδίσει σε σημασία τα επόμενα χρόνια και σίγουρα και λόγω των ενεργειακών ζητημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση ε, ε, αηφορίας και βιωσιμότητας ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα όλων. Αυτό ιδιαίτερα για τις ε, νέες διασυνδέσεις με πετρελαιαγωγούς και αγωγούς φυσικού αερίου ώστε να μπορέσουν να περάσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως νέες εξαρτήσεις όπως για παράδειγμα είναι της Τουρκίας πρέπει να αποφευθούν. Υπό το πολιτικό πρίσμα πιστεύω εγώ ότι η προσέγγιση αρκετών χωρών της Μαύρης Θάλασσας όπως της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να χαιρετήσουμε. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θεμητά ρωσικά συμφέροντα εκεί όπου υπάρχουν σε αυτή την περιφέρεια. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε αυτή η εταιρική σχέση να μην διακυβευτεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι χαιρετίζω τις προσπάθειες ε, της στρατηγικής ε, για τη Μαύρη Θάλασσα που θέλουμε να αποκτήσει νέα όθηση. Είμαι ευγνώμων ε, για την ειλικρινή αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει και δεν θα πρέπει ο ένας υποχρεωτικά να επένει τον άλλον πάντα. Και οι χώρες της περιοχής, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας, του εργατικού δυναμικού και των ενεργειακών πόρων που διαθέτουν. Και βλέπουμε ότι ο Δούναβης εκβάλλει στην ίδια τη Μαύρη Θάλασσα. Ο ευρωπαϊκός ποταμός. Και είναι σημαντικό η συνεργασία των χωρών αυτών στη Μαύρη Θάλασσα να προαχθεί και να λαμβάνουμε και τη μία ε, πτυχή υπόψη και την άλλη. Οι δραστηριότητες των κρατών μελών σε αυτή την περιοχή πρέπει να γίνονται συντονισμένα, να μην ακολουθεί ο καθένα στα δικά του ξεχωριστά συμφέροντα. Και εδώ θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πολυμορφοποίηση, διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα ισχύει αυτό για το πολυμορφικό σχέδιο της, του αγωγού Ναμπούκο, Ναβουχοδονόσορ, αλλά επίσης και για τα εναλλακτικά σχέδια, όπως South Stream, η περιοχή μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Κασπίας και του Καυκάσου, στο Σταυροδρόμι προς την Ασία, Κεντρική Ασία και προς τη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι χαρακτηρίζεται και από παγωμένες σειράξεις και αντιπαραθέσεις. Δεν έχουμε μόνο το θέμα της οικονομίας και της ενέργειας, των ενεργειακών πορών, και της οικονομίας και της σταθερότητας. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας όλο και περισσότερο σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν είναι επόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα αναφέρθηκαν για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για τις ευκαιρίες που διανοίγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Χαίρομαι και με ικανοποιεί ότι βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω προσπάθειες και ανάπτυξη έργου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η ανάπτυξη τώρα της παραμέτρου της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την ίδια τη Μαύρη Θάλασσα ε, έχει ε, κάπως ε, αγνοήσει την πτυχή αυτή. Χαίρομαι για το ότι υπογραμμίζεται τη σημασία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφερική αυτή ανάπτυξη αυτής της περιοχής όχι μόνο για το περιβάλλον και τις μεταφορές αλλά και τις ανθρώπινες επαφές, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση. Είναι σημαντικό να έχουμε ξεχωριστούς στόχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προβλέπουμε κονδύλια υπέρ αυτών, Αλλιώ δεν θα γίνει τίποτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Τικάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η περιοχή του κόσμου και για τις διάφορες εναλλακτικέ διαδρομές για την, την ε, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το... τις κλασικές διαδρομές προς τη Μέση Ανατολή η Ρουμανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εδώ σε σχέση με αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Η Επιτροπή Ήτρε όσον αφορά την στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα λαμβάνει υπόψη είναι αυτά τα πράγματα και είπε και εξ ονόματός μου ότι ο νότιος διάδρομος είναι πολύ σημαντικός για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο Ναμπούκο, Ναβουχοδονόσορ και το δίκτυο προς την Αδριατική θάλασσα ε, και για τη διασύνδεση Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας ή Γεωργίας, Αζερβαϊζάν, Ρουμανίας που έχουν τεράστια σημασία οι παράμετροι αυτοί, αυτές. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θεωρούμε να, ότι ότι ε, πρέπει να εμπλεκόμαστε στην Μαύρη Θάλασσα υπέρ μιας ε, θετικής συνεργασίας και περιφερική συνεργασίας. Η εκπροσώπηση μέσω της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής με την εκπόνηση ενός προγράμματος δράσης για αυτή την περιοχή του κόσμου είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Κάτς διά έχουμε τώρα κυρία Μπλαζέσκου. Έχει το σας ευχαριστώ και πάλι πολύ κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική σημασία της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας του Εύξηνου Πόντου είναι αδιαμφισβήτητη και είναι ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακά, πολιτιστικά, πολιτισμικά, όσον αφορά την ασφάλεια, όσον αφορά τις μεταφορές, όσον αφορά τις γειτονικές σχέσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινοτικής στρατηγικής για την περιοχή, για την περιφέρεια της, του Εύξηνου Πόντου είναι αναγκαιότητα και όχι απλά μια εναλλακτική δυνατότητα, μια εναλλακτική διαδρομή, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια γενικότερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να επιληθούν ε, παγωμένες σειράξεις και αντιπαραθέσεις με την χρήση των ε, δυνατοτήτων αυτής της ζώνης, ιδιαίτερα υπέρ μεγάλης εμβέλειας ε, προγραμμάτων και σχεδίων. Η Ρουμανία είναι υπέρ μιας τέτοιας ευρύτερης στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα και υπέρ μιας στρατηγικής για το Δούναβι μέσα στο πλαίσιο της Μαύρης Θάλασσας. Όλα αυτά καταδεικνύουν με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο πλαίσιο συνεργασίας. Γι' αυτό παρακαλώ κύριε Φίλε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δυνατόν γοργότερα να υιοθετηθεί η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Ο κύριος Πάσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε θα ήθελα πρώτα να πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική πύλη για, προς την Ευρώπη είναι οι λιμένες, τα λιμάνια, μέσω των οποίων οδηγούνται τα εισαγόμενα προϊόντα προς την Ευρώπη ή μέσω των οποίων εξάγονται προς το εξωτερικό τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η σημασία των λιμένων είναι τεράστια και αυτό όχι μόνο στις ε, παράκτιες περιοχές αλλά και εσωτερικά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα λιμάνια των ε, ποταμών μας όπως του Δούναβη για παράδειγμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οικονομικά έχει τεράστια σημασία να μπορούμε να αναφερθούμε στα έγγραφα τα οποία πρέπει να συντονίζουμε όσον αφορά τη στρατηγική μας για το Δούναβη και για τον Εύξηνο Πόντο. Στρατηγικά στοιχεία που πρέπει να συντονίζονται όσον αφορά τις περιφέρειες αυτές Δούναβη και Εύξηνο Πόντο, ώστε να υπάρξουν συνέργειες, ώστε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τον φυσικό πλούτο και το δυναμικό, ώστε να είναι μεγαλύτερες οι δυνατότητες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία αυτά τα οποία αφορούν και τον πλούτο, τον ορυκτό ε, και ότι ε, έχουμε 150 εκατομμύρια ε, καταναλωτές σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας έχει τεράστια σημασία. Η διαπεριφερειακή συνεργασία πρέπει να τύχει μεγαλύτερης εκμετάλλευσης ως μοχλός, ως στοιχείο, ώστε στην πολιτική γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ένα ε, ζίδωρο στοιχείο. Όμως ε, έχουμε μια ιδιαίτερα θα έλεγα χαμηλού προφίλ εκπροσώπηση όσον αφορά την ε, ενδυνάμωση της, γειτονικής, της πολιτικής γειτονίας. Η περιφερειακή αυτή συνεργασία πρέπει να προαχθεί με τη δημιουργία και υιοθέτηση μιας αυθεντικής στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκκινεί από τις συνέργειες στον εύξηνο πόντο λαμβάνοντας υπόψη και αφομοιώνοντας και τις πτυχές της συνεργασίας για την λεκάνη του Δούναβη. Ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μία ερώτηση θα, είχα, θα ήθελα να διατυπώσω στην ε, ε, εξέλιξη, στην ανάπτυξη του ε, διαδρόμου αυτού δεν υπάρχει κάποιο κονδύλιο που να προβλέπεται ενώ υπάρχουν κονδύλια για άλλες δράσεις ε- από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια συμφωνία, ένα υπόμνημα, ένα memorandum για τη διάνοιξη αυτών των διαδρόμων. Παρακαλούμε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κονδύλια τα οποία θα δεσμεύσει υπέρ αυτών των διαδρόμων, ώστε οι διάδρομοι της Μαύρης Θάλασσας να μπορέσουν να ανοίξουν, να διανοηθούν και να λειτουργήσουν, όπως και στη Βαλτική ή στη Μεσόγειο χρηματοδοτούνται τέτοιοι διάδρομοι. Δεν υπάρχει κάποια συνολική σφαιρική συμφωνία όσον αφορά την εκμετάλλευση της αλίας για παράδειγμα μέσω συνέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προαγάγει τον περιφερειακό διάλογο για μια τέτοια κοινή στρατηγική στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου. Να λάβει υπόψη και τη συμμετοχή των άλλων γειτονικών των όμορων χωρών. Σας ευχαριστούμε κυρία Τικάου. Τώρα η διαδικασία Catch the Eye που ολοκληρώθηκε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σε σχέση με την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Φιούλε. Παρακαλώ. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την σύντομη, όμως πάρα πολύ εμπνευσμένη ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά την συνεργειακή στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα. Εγώ, εγώ κρατώ την πεποίθηση ότι από κοινού θα πετύχουμε όσον αφορά την συνέργεια, όσον αφορά την ευρύτερη συνεργασία με την περιοχή αυτή, όσον αφορά την ε, ολοκληρωμένη μας πολιτική για τη θάλασσα, αλλά και την στρατηγία των τον Θα μπορέσουμε έτσι τελικά να φτάσουμε εις αυτήν την ε, φάση όπως την περιέγραψε ο τελευταίος αγορητής αλλά και η συνάδελφος Μαρία Δεμανάκη ξεκίνησε αυτή τη ε, ε, διαδικασία όπως ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια διαδικασία, μια διαχειριστική διάταξη και να φτάσουμε σε μια διαχείριση των αλληλευτικών πόρων που να είναι αηφόρος. Στο Βουκουρέστι θα γίνει σχετική διάσκεψη, όπως γνωρίζετε, τον Νοέμβριο φέτος. Και έτσι θα αυξηθούν οι δυνατότητες για συνεργασία. Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σχετικές προκλήσεις. Την πολιτική, για την ασφάλεια, την θεράσια πολιτική και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αναβάλλονται της εμπιστοσύνης όσον αφορά τη μαύρη θάλασσα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανθεωρήσει την πολιτική της. Θα πρέπει να εξετάσει την οικονομική διάσταση και να δει πώς είναι δυνατόν να πετύχει τους στόχους της. Και βέβαια εμείς υπολογίζουμε στην ε, Συμπάρξη του Ευρωβουλίου περιμένω πώς και πώς τις συστάσεις. Γι' αυτό, πέστε μας, πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στην πολιτική που έχουμε γράψει για τη Μαύρη Θάλασσα και ταυτόχρονα να δουλεύουμε σκληρά όσον αφορά τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε προναφέρει. Άκουσα και τίποτε ορισμένοι εξημών. για την έχει ασφάλεια. για την συνεργασία, τον δημοκρατισμό όσον αφορά τη στρατηγική αυτή. Κοιτάξτε, δουλεύουμε σκληρά για όλα αυτά και προανέφερα ότι αφορά όσον αφορά την συνεργασία μας προς Ανατολάς. Και έτσι Προσπαθούμε να ακουστεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια εκείνη. Και τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη συζήτησή μας είναι το εξή. Και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Πολλοί ζητούν μια τέτοια στρατηγική και ένα θεσμικό πλαίσιο. Όμως, τους έχω καλέσει να έρθουν και να μας παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πού να τα προσθέσουμε στην ασκούμενη πολιτική, να μπορέσουμε έτσι να φτιάξουμε κάποιους πυλώνες, κάποια δομή. Να σας πω την αλήθεια, όλοι αυτοί μπορούσαν να προσφέρουν κάποια πρόταση που να στέκει. Και έτσι προχωρούμε προς αυτή την εταιρική σχέση προς Ανατολάς και αστεριώνουμε μια τέτοια σχέση με τους εταίρους μας σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου. Και όλο ένα και περισσότερο θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία και και να εξασφαλίσουμε να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Είμαστε όλοι αρσατοί. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε φίλε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ Αζερβαϊτζάν και ΕΕ Αρμενίας. Η μία έκθεση έχει συντάκτη την κυρία Γέτεν Μέκη για τις διαπραγματεύσεις ε, για την συμφωνία σύνδεσης